Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να σας διακόψω. Διότι θα πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Καλησπέρα σας. Καλωσορίζω όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής ΙΤΡΕ Βιομηχανίας. Είναι η πρώτη πλήρης τακτική συνεδρίασή μας όχι τακτική, βασικά έκτακτη είναι γιατί είναι συνεδρίαση ακρόασης του Οριστέντος Επιτρόπου. Καλωσορίζουμε ορίζουμε και του συναδέλφου των Επιτροπών ΕΝΒΙ, και Μεταφορών που συμμετέχουν ή συμμετείχαν μάλλον στην ακρόαση του κυρίου Αντώνιο Ταγιάννη, πρώην Αντιπροέδρου Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2009. Σας καλωσορίζω όλους λοιπόν. Και επιτρέψτε μου όλος ιδιαίτερος να καλωσορίσω θερμότατα τον κύριο Νέλη Φερότσι που είναι οριστής επίτροπος βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας. Πάρα πολύ σημαντική αυτή γιατί είναι το σημερινό μας θέμα η βιομηχανία καθώς και η επιχειρηματικότης. Θα είναι το θέμα που θα κυριαρχήσει σήμερα στη συζήτησή μας. Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ και τους Γερμανούς συναδέλφους εμπαρόδο και τους Ολλανδούς όμως. Μπράβο σας. Επάξια εκπροσωπήσατε σύνολη την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχουμε και εμείς σε αυτή τη νίκη σας. Μπράβο. Um, like to give... Θα ήθελα επίσης ε, αρχικά να σας κάνω κάποια σχόλια. Πρώτον, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Κοινοβούλιο αξιολογεί όλους τους οριστένες επιτρόπους, βάσει των γενικών τους ικανοτήτων ε, της Ευρωπαϊκής Δέσμευσης και προσωπικής ανεξαρτησίας ως κριτήρια. Επίσης αξιολογείται και η γνώση σχετικά με το χαρτοφυλάκιο που θα αναλάβουν και τα επικοινωνιακά τους ε, προσόντα. Ε, αυτά τα λέει ο κανονισμός μας και είναι και πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά... Ε, ε πριν τη συνεδρίασή μας λοιπόν ε, ορίστηκε ο κύριος Νέλη Φερότσι και απάντησε γραπτός σε ένα ερωτηματολόγιο που διατίθεται σε όλες τις γλώσσες ε, των μελών της Επιτροπής μας και των υπολείπων επιτροπών που συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή. Θα ήθελα να προσθέσω το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων μας επίσης πάρα πολύ σημαντικό ε, ή τις παρούς συνεδρίες. Πρώτον, θα δώσω το λόγο στον κύριο Νέλη Φερότσι για μια εισαγωγική τοποθέτηση που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 λεπτά. Κύριε Πρέσβη, αν μου επιτρέπετε, στο ζητήσω. Και μετά την εισαγωγή αυτή θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και απαντήσεις διάρκειας 35 λεπτών. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι ορίσουμε τον κύριο Νέλη Φερότσι ε, μόνο για λίγους μήνες μέχρι να αναλάβει η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή το φθινόπωρο. Δηλαδή είναι έτσι μια απλουστευμένη ακρόαση για να το πω έτσι. Και η κατάσταση θα είναι πολύ διαφορετική το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο στις άλλες ακρόασεις. Αν υπάρξει ακρόαση στην Επιτροπή μας που θα υπάρξει, γιατί τέσσερις σίγουρα θα έχουμε. Λοιπόν, έλεγα 35 λεπτά στην αρχή, ερωτήσεις. Ένας εκπρόσωπος κάθε πολιτικής ομάδας, αρχικά, οκτώ δηλαδή, επικεφαλής των πολιτικών ομάδων στην Επιτροπή μας. Και σύμφωνα με τη διαδικασία την αρχή του πινκ-πονγκ, ερώτηση-απάντηση αμέσως. Πολύ σύντομη ερώτηση και στη συνέχεια αρκετά σύντομη απάντηση του κυρίου Πρέσβη. Συνολικά λοιπόν, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το τρίλεπτο ερώτηση και απάντηση. Ή δυνατόν ένα λεπτό η ερώτηση και δύο λεπτά η απάντηση. Αν μπορείτε και πιο σύντομα ακόμα καλύτερα για να έχει περισσότερο χρόνο ο κύριος να απαντήσει στην ερώτησή σας. Και αν έχουμε αρκετό χρόνο, ίσως να προσθέσουμε και δύο επιπλέον ερωτήσεις. Οι συνάδελφοί μας των Επιτροπών Περιβάλλοντος Εσωτερικής Αγοράς και Μεταφορών Δεν θα κάνουν τώρα ερωτήσεις, αλλά στην κανονική διαδικασία μας, το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, θα έχετε την ευκαιρία. Όπως άλλωστε έγινε και με την περίπτωση του κυρίου Ταγιάννη, αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη δική του ακρόαση, το Σεπτέμβριο του 2009. Λοιπόν, στο τέλος συνεδρίασής μας, ο Υιβιστής Επίτροπος θα έχει την ευκαιρία να κάνει μια σύντομη καταληκτική δήλωση. Και παρακαλώ ιδίως τα νέα μέλη του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής να τηρούμε ε, ε, αυτά και να μην μιλάμε πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί πρέπει να μεταφραστούν και σε όλες τις γλώσσες. Όταν μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα δεν σας προλαβαίνουν οι διερμηνείς. Και δεν μπορούν να μεταφράσουν σωστά αυτά που λέτε. Παρακαλώ έτσι, σκεφτείτε το αυτό. Άρχεται λοιπόν η ακρόαση. Νομίζω ότι καταλάβαμε όλοι τους κανόνες. Αγαπητοί φίλοι, πάμε. Κύριε υποψήφιο επίτροπε, παρακαλώ έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, ε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, Κυρίες και κύριοι, θέλω καταρχάς να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο και καλή δουλειά με επίγνωση ότι βρίσκεται, βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μιας θητείας που είναι αποφασιστική για το μέλλον της Ευρώπης. Όπως κάποιοι από εσά γνωρίζετε, η ευρωπαϊκή δέσμευση ήταν καθοδηγητήρια κατά μία της, ε, της προηγούμενης επαγγελματικής μου καριέρα. Πολλές φορές είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω τις εξελίξεις του ευρωπαϊκού εγχειρήματος από άλλη θέση, ως εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης ιδίως ε, στην τελευταία περίοδο ως μόνιμος αντιπρόσωπος της Ιταλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θέση που εγκατέλειψα πριν από ένα χρόνο μόνο. Σήμερα παρίσταμε ενώπιόν σας στην ακρόαση αυτή με διαφορετικό ένδυμα ως ε, οριστής επίτροπος με ευθύνη την επιχειρηματικότητα και τη βιομηχανία. Έχω πλήρη επίγνωση του νέου ρόλου και των νέων ευθυνών μου. Και τούτο και του τι σημαίνει κάτι τέτοιο ως προς την ανεξαρτησία και την αυτονομία μου. Να προσθέσω επίσης ότι έχω επίγνωση και των ευθυνών μου έναντι του Κοινοβουλίου. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να εκφράσω εξ αρχής την πλήρη διαθεσιμότητά μου αν με επικυρωθώ στη θέση αυτή, να συνεργαστώ μαζί σας σε έναν μόνιμο ανοιχτό, νόμιμο και διάφανο διάλογο μαζί σας. Τέλος, το είπε και ο πρόεδρος, το επαναλαμβάνω και εγώ, η εντολή είναι, η θητεία είναι μια θητεία βραχία μέχρι την ολοκλήρωση της τωρινής επιτροπής. Ωστόσο, ε, θέλω να τιμήσω την περίοδο αυτή με πνεύμα συνέχεια σε σχέση με το έργο του προκατοχού μου κ. Ταγιάννη, που ευχαριστώ για όσα έκανε στην ε, θέση που είχε ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Παρελθόν. Κύριε Πρόεδρε, η κρίση που δημιουργήθηκε ως κρίση δημοσίου χρέους έπληξε και την πραγματική οικονομία. Φέτος η βιομηχανία έχασε 4 εκατομμύρια θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και 350 δις επενδύσεων. Τα μέτρα που υιοθετήθηκαν τα χρόνια αυτά για να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των δημοσίων του προϋπολογισμού ε, επέτρεψαν να σταθεροποιηθεί η Ευρωζώνη, ωστόσο είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία. Υπάρχει μια πλήρης επίγνωση σήμερα ότι οι προτεραιότητε στην Ευρωπαϊκή Μερίσια Διάταξη θα πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη και τη μάχη κατά της ανεργία, ιδίω τη ανεργία των νέων. Από αυτή την οπτική η βιομηχανία και η επιχείρηση πρέπει να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από την ικανότητά της να αναλάβει εκ νέου την ηγεσία στον ε, βιομηχανικό τομέα. Άρα απαιτείται κοινή δέσμευση που θα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Μηχανία να συμβάλλει απόφαση περισσότερο στην βιώσιμη ανάπτυξη και στην αύξηση των θέσεων εργασία. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνει μέσω ενό φιλόδοξου προγράμματο ανάκτηση τη ανταγωνιστικότητα με επίγνωση ότι η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα δεν είναι ασύμβατες αρχές αλλά μπορούν να ενισχύσουν η μία την άλλη και αμοιβαία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του περασμένου Μαρτίου κατέγραψε όλα αυτά. Η Ευρώπη προσβλέπει με νέα επίγνωση και με νέα στάση την πραγματική οικονομία. Δημιουργείται μια ευρεία συνένεση και την ανάγκη να αναθεωρηθούν οι προτεραιότητες σε μια ευρωπαϊκή μερίσια διάταξη που μέχρι τώρα έδινε στόχο, έθετε προτεραιότητα στην δημοσιονομική πειθαρχία και στηριζόταν σε μακροοικονομικές διαστάσεις κυρίως, αφήνοντας λίγο χώρο στη μικροοικονομική διάσταση που εξορισμού είναι πιο κοντά στις επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία. Είναι σημαντικό από αυτή την άποψη το ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο Μάρτιο πάντα αναγνώρισε τον κεντρικό χαρακτήρα της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης που θεωρήθηκε ως κινητήρα στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Οι προτάσεις που έκανε η Επιτροπή με την ανακοίνωσή της του περασμένου Ιανουαρίου ήταν, αποτέλεσμα, ε, ήταν και στη βάση αυτών των θέσεων. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θετήθηκε από τους προκατόχους στην Επιτροπή αυτή με την εξαιρετική έκθεση Μπουτικόφερ για το θέμα αυτό. Ο, η σύνοδος κορυφής λοιπόν του περασμένου Μαρτίου έδειξε μια σαφή πορεία. Ένα από τα επιτεύγματα της πορείας αυτής ήταν το αίτημα που απευθύνθηκε προς την Επιτροπή να προετοιμάσει ένα roadmap με λεπτομέρειες που θα καθορίζει τις πρωτοβουλίες και τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτός ο οδικός χάρτης, το roadmap, θα υποβληθεί από την επόμενη επιτροπή στο ξεκίνημα του 2015. Πρόθεσή μου είναι ωστόσο να προτείνω στο, στο Κολέγιο των Επιτρόπων να ξεκινήσει ήδη την προπαρασκευαστική δουλειά. Και εύχομαι και το Κοινοβούλιο να συμβάλλει στο εγχείρημα αυτό με τον τρόπο που θα θεωρήσει πλέον σκόπιμο. Με βάση τις ενδείξεις που δόθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο δικός χάρτης θα στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες. Πρώτον, πρόσβαση στην αγορά στις αγορές, τόσο την εσωτερική αγορά όσο και τις διεθνείς αγορές. Από την πρώτη οπτική αναγνωρίζεται ότι τη σημαντική πρόοδος που έχει γίνει μέχρι τώρα στην νέα αγορά που πρέπει ωστόσο να συμπληρωθεί με επιπλέον μέτρα για την ε, άρση των υπόλοιπων εμποδίων που συνιστούν εμπόδια στην ανταγωνιστικότητα και την ε, μεγάλη διάσταση των επιχειρήσεων. Παράλληλα θα πρέπει να προωθηθεί μια αποτελεσματική στρατηγική διεθνοποίησης και πρόσβαση στην αγορά των τρίτων χωρών από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ένα σημαντικό ρόλο στην άποψη αυτή, στη θέση αυτή θα παίξουν οι συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου που συνάπτει, ή διαπραγματεύεται ενέσου με κάποιους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους. Θα διασφαλίσω ότι στις διαπραγματεύσεις αυτές αξιοποιούνται οι δυνατότητες για καλύτερη πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στι αγορές των τρίτων χωρών και ταυτόχρονα θα λαμβάνονται υπόψη και τα αμυντικά συμφέροντα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Ο δεύτερος άξονας είναι η πρόσβαση στους πόρους. Πρόθεση της Επιτροπής είναι να θέσει στη διάθεση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων επιχειρήσεων κατάλληλα εργαλεία για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην ε, ε, εμπορική πίστη. Θα μιλήσω αργότερα για το πρόγραμμα COSME και Horizon 2020, αλλά και πρόσβαση σε σταθερή αξιόπιστη βάση και για τις ε, πρώτε ύλε που είναι αναγκαίε για την παραγωγική δραστηριότητα στην Ευρώπη και κυρίω στι πηγέ ενέργεια. Για το τελευταίο αυτό θέμα, που είναι κρίσιμο, την ενέργεια δηλαδή, Θυμίζω ότι η Επιτροπή θέλει να δραστηριοποιηθεί σε πολλά μέτωπα για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας συμπληρώνοντας την εσωτερική αγορά ενέργειας και βελτιώνοντας την, αποτελεσ... την ενεργειακή αποτελεσματικότητα μειώνοντας ταυτόχρονα την εξάρτηση από το εξωτερικό. Εν τέλει, η Επιτροπή δεσμεύεται να προωθήσει την διαθεσιμότητα επαγγελματικών προσωπικότητων με ικανότητα για τις επιχειρήσεις και την ε, επιχειρηματικότητα με το πρόγραμμα Εράσμους για νέους επιχειρηματίες πληροφορίες αναδεικνύοντας τα συστήματα διπλής εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχει δώσει πολύ καλά αποτελέσματα σε κάποια κράτη-μέλη. Ο τρίτος άξονας είναι η υποστήριξη καινοτομία. Καινοτομία που θα πρέπει να παίξει ουσιώδη ρόλο για τη βελτίωση της αγωνιστικότητας. Ήδη ξεκίνησαν πολλές πρωτοβουλίες με, στόχο, με τον στόχο αυτό και χρηματοδοτούνται ε, ιδίως μέσω του προγράμματος Horizon 2020. Σημαντική διάσταση που αξίζει να αναφερθεί είναι οι τεχνολογίες κλειδιά που μαζί με τις πράσινες τεχνολογίες θα είναι οι κύριοι κινητήρες καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας ε, στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Να υπογραμμίσω επίσης και το σημαντικό ρόλο που παίζουν τα οι διαφορετικοί πόροι και οι περιφερειακοί κυρίως πόροι για την ε, περίπου ύψου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ που είναι στη διάθεση των ευρωπαϊκών περιφερειών για να τις επιτρέψουν να αναπτύξουν οι ίδιες βιομηχανική καινοτομία. Ο τέταρτο άξονα, εξίσου σημαντικό με τι προηγούμενες, ίσως και περισσότερο, έχει να κάνει με την ποιότητα της νομοθεσία. Στο πλαίσιο των δράσεων που έχει ξεκινήσει η Επιτροπή με το REFIT, δέσμευση, υπάρχει δέσμευση από πλευρά μου στο πλαίσιο της ιδίας μου να χρησιμοποιήσω τα εργαλεία αυτά που θα μας που θα μας επιτρέψουν να μειώσουμε την υπερβολική νομοθεσία και να μειώσουμε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων. Ιδίω σκέφτομαι την μελέτη αντικτύπου, την αξιολόγηση αντικτύπου, το εργαλείο του Competitiveness Prouting, την αξιολόγηση των σωρευτικών κοστών στο στα, στις δοκιμές αντικτύπου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο από την υφιστάμενη ή μελλοντική ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και για τις εθνικές νομοθεσίες όπως ήδη ανέφερε πάλι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Μάρτιο. Τα εργαλεία αυτά πρόθεσή μου είναι να τα υλοποιήσω μέσω της αρχής του mainstreaming, δηλαδή να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι ο στόχος ανταγωνιστικότητας θα λαμβάνεται συστηματικά υπόψη στην επεξεργασία και έγκριση ευρωπαϊκών νομοθετικών κειμένων. Μια αποτελεσματική στρατηγική βιομηχανική αναγέννηση θα πρέπει να εμπλέκει αναγκαστικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συμβάλλουν κατά 80% σήμερα στις νέες θέσει εργασίας, δίνοντα θέσει εργασίας σε 87.000 άτομα 27 ε, εκατομμύρια άτομα ενώ βελτιώνουν την ε, οικονομική δραστηριότητα. Η Επιτροπή τώρα έχει νέα σημαντικότερα εργαλεία για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θυμίζω το πρόγραμμα COSME και κάποιες διαστάσεις του προγράμματος Horizon. Θα μιλήσω λεπτομερέστερα για τα θέματα αυτά αν τεθούν ερωτήσεις για τον τρόπο λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών. Να θυμίσω εν τέλει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι η Επιτροπή θέλει να ενεργοποιήσει απόλυτα ε, την νομοθεσία, το Small Business Act και να ενημερώσει για την ε, εφαρμογή και υλοποίηση του Small Business Act με στόχο να εξετάσει τις πιθανότητες μελλοντικών ε, εξελίξεων στον τομέα αυτό. Θα μπορούσατε να συνοψίσετε με λίγες προτάσεις ακόμα κύριε Πρέσβη. Βεβαίως, δίκιο έχετε. Δύο λόγια για να πω ότι η Επιτροπή δεσμεύεται να αναπτύξει ειδικού προπολογισμού για όριμους τομείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας όπου έχουν ξεκινήσει ήδη μελέτες, ε, χάλιβας, ε, κατασκευαστικές ε, δραστηριότητες και να τονίσω τα προγράμματα που έχουμε ξεκινήσει στο θέμα του διαστήματος. Κοπέρνικος και Γκαλιλαίο ιδίω. Επίσης, πρόεδρε, να κλείσω θυμίζοντας ότι λόγω της οικονομικής κρίσης οι Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν ότι η Ένωση είναι μακριά από αυτούς και δεν ενδιαφέρεται για τα προβλήματα και τις ενθυχίες τους. Τα ευρωπαϊκά όργανα πρέπει να εκμεταλλευτούν όσο καλύτερα γίνεται την ε, υποστήριξη της κοινή γνώμης των κρατών μελών για το ευρωπαϊκό εγχείρημα και πιστεύω πραγματικά ότι η ευρωπαϊκή μερίσια διάταξη ε, με έμφαση στην ευρωπαϊκή οικονομία και την ανταγωνιστικότητα των μηχανιών θα συμβάλλει στις θέσεις εργασίας και θα φέρει το ευρωπαϊκό εγχείρημα κοντά στους πολίτες. Εάν επιβεβαιώσετε την τοποθέτησή μου την Επιτροπή, ως Επιτρόπο Βιβανίας πρόθεσή μου είναι να συνεργαστώ με αυτό το στόχο υπόψη και έχω εμπιστοσύνη στο ότι μπορώ να συνεργαστώ απόλυτα μαζί σας στην ε, επεξεργασία της πολιτικής αυτής. Είμαι ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σα. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη. Ερωτήσεις λοιπόν τώρα από τους συντονιστές καταρχάς. Κάρινς, τρία λεπτά ερώτηση και απάντηση μαζί. Καλό θα ήταν ε, να μην ξεπεράσετε τον λεπτό στην ερώτησή σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φερότσι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είστε δεσμευμένο υπέρ τη ευρωπαϊκή ιδέα, όπω φαίνεται ξεκάθαρα από το βιογραφικό σα. Στην Επιτροπή μα ε, όμω ε, η λέξη κλειδί είναι ανταγωνιστικότητα. Πώ μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Ω προσωρινό επιτρόπο που παίρνετε τα από τον κύριο Ταγιάννη, θα έχετε λίγου μήνε μόνο στη διάθεσή σα και μπορείτε είτε να ακολουθήσετε το ίδιο μονοπάτι, είτε να προσπαθήσετε να προωθήσετε κάποιε διαφορετικέ θα ήθελα να σχολιάσετε ε, τι είναι αυτό που εσείς θα θέλατε να κάνετε και πώς ε, θα προσεγγίσετε τους ε, ομολόγους σας επιτρόπους στο θέμα της ανταγωνιστικότητας αλλά και δύο σε δύο τομείς. Ο πρώτος είναι η ενέργεια. Αναφερθήκατε και στην ενέργεια. Πρέπει να αυξήσουμε την απόδοση γίνεται λόγος για αύξηση του κομματιού του μεριδίου της, ε, των ανανεώσιμων ETS, εμπορία εκπομπών. Πώς μπορείτε κόστος και ανταγωνιστικότητα έναντι ενεργειακών στόχων να εξισορροπήσετε αυτή την εξίσωση. Απάτηση. Γνωρίζω πολύ καλά το χρονοδιάγραμμα, ξέρω πόσο θα διαρκέσει η θητεία μου και ουσιαστικά η ιδέα μου είναι να ακολουθήσω το πνεύμα της συνέχειας, δηλαδή να ακολουθήσω στα βήματα του προκατόχου μου. Η ανταγωνιστικότητα θα είναι σίγουρα ε, κλειδί, ε, θα μας εμπνεύσει, θα εμπνεύσει τη δράση μου στην Επιτροπή. Δύο είναι τα βασικά μου καθήκοντα. Ένα, προνέφερα, είναι η εκπόνηση του οδικού χάρτη που θα υποβληθεί επισήμω από την ε, επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ήδη επεξεργαζόμαστε ορισμένου τόμου προτεραιότητα. Μεταξύ αυτών, σε μεγάλη, σε ψηλή θέση θα είναι η πρόσβαση στου ε, πόρου για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όταν ε, λέω πρόσβαση στους πόρους, τι εννοώ το ανέφερα βέβαια συντομία, μιλώ στην για πρόσβαση σε πρώτες ύλε, αλλά και σε ενέργεια σε προσιτές τιμές. Εύκολο δεν θα είναι, είναι ένα συλλογικό καθήκον, αφορά όλους τους επιτρόπους, σίγουρα όμως ε, θα είναι δική μου ευθύνη συγκεκριμένα να επεξεργαστώ τις ε, συνιστώσεις ε, τις ενεργειακές ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα. Αναφερθήκατε ε, και σε άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τελικά το κόστος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ETS δηλαδή σύστημα εμπορίας και θέλω να σας πω ότι δεν ε, κάνει τις προτάσεις της μόνο η Κομισιόν, εγκρίνει και το Συμβούλιο όπως ε, το καθεστώς για τις ε, επιχειρήσεις έντασης ενέργειας θα ισχύσει λοιπόν και στο μέλλον και αυτό νομίζω ότι απαντά κάπου σε ανησυχία σας. Ευχαριστώ, διακόπτει ο Πρόεδρος. Well, two, sentences at the end, if you wish. No, uh... Για να ολοκληρώσω, ε, τα υπόλοιπα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα της ε, Επιτροπής, ενεργειακή απόδοση, ασφάλεια της ενέργειας και σύντομα δυνάμει μιας αξιολόγησης για την ε, υλοποίηση της σχετικής οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση θα παρουσιάσει νέους στόχους η Κομισιόν και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα, αλλά να λάβουμε ταυτόχρονα υπόψη τον ενεργειακό παράγοντα. Ευχαριστώ. S&D Νίκα. Κύριε είναι Προφανές ότι είναι πολύ μικρή εναπομείνασα περίοδος της ευρωπαϊκή Επιτροπής. Δεν μπορεί κανείς να ξεκινήσει μεγάλες ε, πρωτοβουλίες για μεγάλες πολιτικές. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόζεται σωστά και αποτελεσματικά η κείμενη νομοθεσία και να συνεχίσει. Θα μπορούσατε να μας πείτε με λεπτομέρειες ποιες θα ήταν οι δικές σας προτεραιότητες ε, για την εφαρμογή αυτών έχετε συζητήσει με τον προκάτοχό σας για τα βασικότερα στοιχεία που θα πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας και μπορείτε λίγο να μας αναφέρετε ποια θα είναι αυτά. Ευχαριστώ. Uh, Μάλιστα. Πρώτη μου δέσμευση για αυτή τη θητεία μου θα ήταν να εξασφαλίσω μία ομαλή Ε, συνέχιση της εξέτασης των διαφόρων φακέλων που έχουν δρομολογηθεί στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Και εδώ σκέφτομαι τρία νομοθετικά μέτρα που εξετάζονται ήδη και από το Συμβούλιο αλλά και από το Κοινοβούλιο. Το πρώτο είναι η δέσμη ή το πακέτο για την επιποπτεία των αγορών και την ασφάλεια των προϊόντων. Το δεύτερο είναι ο κανονισμός για την καταχώρηση οχημάτων και το τρίτο είναι ε, το λεγόμενο ηλεκτρονικό τηλεφώνημα ή κόλ, επίσης ε, κανονισμός. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουν οριμάσει προς έγκριση κατά τη διάρκεια της αιτίας της παρούσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτά τα τρία θέματα. Και σε ό,τι αφορά ε, τις ανταλλαγές που είχα και τις επαφές με τον κύριο Επίτροπο, συγγνώμη, τώρα Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Ταγιάννη, βεβαίως είχαμε ανταλλαγή απόψεων πριν αναλάβω αυτή την υποψηφιότητα και όσα έχουμε πει και όσα θα σας πω και σε όσα θα απαντήσω είναι πάντα σε συνεννόηση μαζί του με τη Γενική του Διεύθυνση και το ιδιαίτερο γραφείο του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέσβη. Επόμενος ομιλητής. Κάποιος από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ο συνάδελφος Ρουμπάρσεκ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, πολωνικά. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στο εξή θέμα. Ε, και εγώ για την ενέργεια ενδιαφέρομαι και για το υψηλό κόστος της ενέργειας. Αυτό που μας ενδιαφέρει να μειωθεί η τιμή της ενέργειας διότι όταν είναι ακριβή ενέργεια ε, φεύγουν ε, οι βιομηχανίες από την Ευρώπη κλείνουν τα εργοστάσια, ιδιαίτερα χαλιβουργίες και αυτοκίνητο βιομηχανίες. Δεύτερον, μελέτη αντικτύπου. Αναφερθήκατε σε αυτό. Εδώ και χρόνια γνωρίζουμε ότι οι μελέτες αντικτύπου είναι κάτι το αρνητικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μιλώ πάντα για τις ρυθμίσεις και το φόρτο. Εν ώψη όλων αυτών, εσείς τι προτίθεστε να πράξετε έτσι ώστε να ε, εξαφανιστεί αυτή η αρνητική επίπτωση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Η νομοθεσία θα πρέπει να είναι πιο φιλική προς τις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Για το κόστος της ενέργειας και πώς αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα βιομηχανίες με ένταση ενέργειας, ενεργοβόρες ιδιαίτερα. Σας είπα για το καθεστώς αυτό ότι θα διατηρηθεί και στο μέλλον για αυτό που διέπει τις ενεργοβόρες ε, επιχειρήσεις που μεταγκαθίστανται, το λεγόμενο carbon leakage. Ε, ξέρουμε ότι υπάρχει ιδιαίτερη επιβάρυνση για αυτές τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Ενδέχεται ε, να εγκριθούν νέοι όχι ε, για ε, τα αέρια του θερμοκηπίου. Τον Οκτώβριο θα το συζητήσει αυτό το θέμα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το επόμενο λοιπόν καθεστώς εμπορίας εκπομπών ρήπων ETS θα καλύψει προσεκτικά τους τομείς και θα τους εξαιρεί ε, από το ETS. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επιπλέον δεσμεύομαι και δεσμεύω και τις υπηρεσίε ότι θα παρακολουθούμε στενά την προετοιμασία της νομοθεσίας που θα χρειαστεί για να εφαρμοστούν οι νέοι στόχοι εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Έτσι ώστε να αποφύγουμε ε, άχρηστες επιβαρύνσεις και περιττό κόστος για τις επιχειρήσεις. Βέβαια παραμένει ο στόχος μείωσης του ε, διοξιδίου του άνθρακα. Για τις μελέτες αντικτύπου και τι έχει γίνει, θα μπορούσε να γίνει περαιτέρω για να μειωθεί ε, το υπερβολικό άχθος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ προσελωμένος σε αυτή την προσπάθεια. Ε, θα χρησιμοποιήσω ό,τι δυνατότητα έχουμε, αλλά στα πλαίσια της αναθεώρησης του Small Business Act που εξήγηλα, με έγγραφο, για, για δημόσια διαβούλευση θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, αλλά αυτό είναι θέμα της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ενδεχόμενο υποβολής νομοθεσίας για την υλοποίηση ειδικών στόχων για τη μείωση του κόστους για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Και μείωση και των χρόνων αναδιαδότησης Ευχαριστώ. Συγγνώμη, έληξε ο χρόνος σας, ο Πρόεδρος. Ο συνάδελφος Ντεμπάκερ από τους Φιλελευθέρους, παρακαλώ. Ευχαριστώ να καλησπέρισω τον κύριο Φερότσι. Έχω δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι ότι του επόμενου μήνε και δύο-τρία χρόνια που ακολουθούν θα μιλάμε για καινοτομία και ανταγωνιστικότητα κυρίω Για να εφαρμοστεί βιομηχανική πολιτική που σχεδίασε ο προκατοχό σα, θα χρειαστεί και η βοήθεια από τα κράτη-μέλη που και αυτά θα πρέπει να υλοποιήσουν δομικέ δραστηριοτικές μεταρρυθμίσει ε, σε ό,τι αφορά την ετήσια έρευνα για την απασχόληση, το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Στου επόμενου μήνε. τι δράσει μπορείτε να αναλάβετε ώστε η υλοποίηση ε, που εδώ έχουμε πρόβλημα, 20% μόνο των στόχων έχουν επιτυχθεί επιτευχθεί, πώς θα γίνει τους επόμενους μήνες ε, να μεγαλώσει αυτό το ποσοστό για να προετοιμάσουμε τον επόμενο κύκλο. Δεύτερο ερώτημα για την υγειονομική περίθλαψη και την καινοτομία. Πολλές εψηλών, να δραστηριοποιούνται στον τομέα των φαρμάκων, βιοτεχνολογίας, αλλά αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα. Έχουμε όμως και γύρανση του πληθυσμού. Πώς εδώ μπορείτε τη στήριξη για ΜΜΕ, την καινοτομία, να τα συσχετίσετε και πώς μπορούν να βοηθήσουν και τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν δηλαδή τον προπολογισμό υγείας για να προωθήσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση. Απάντηση για το πρώτο σας ερώτημα κύριε Ντεμπάκερ, ε, αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι πολλά πρέπει να γίνουν από τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά ε, τη δημιουργία ενός ε, περιβάλλοντος που θα είναι φιλικό για την επιχειρηματικότητα και για τις, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης ε, στηρίζω τα μάλλα και την ιδέα σας για την καλύτερη ενσωμάτωση ε, των ε, πολύ μικρών επιχειρήσεων και των συμφερόντων τους και στις συστάσεις αναχώρα και στην πολιτική του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αυτό το μήνυμα θα το μεταφέρω βέβαια μάλλον στον διάδοχό μου, γιατί νομίζω ότι για να πετύχουμε αυτό το στόχο Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για τον Επίτροπο που θα είναι αρμόδιος για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη στήριξη τους για την τόνωση της καινοτομίας, νομίζω ότι έχουμε πολλά εργαλεία. Ε, το κόσμε ε, δεν το προανέφερα, αλλά είστε, να είστε βέβαιοι ότι το κόσμε ε, που είναι διάδοχος του CIP είναι για την του μέσου για την καινοτομία για τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο και θα τονώσει μεταξύ άλλων την καινοτομία. Κάτι άλλο σημαντικό που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ορίζον 2020, το νέο πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και καινοτομία. Αυτό το πρόγραμμα επικεντρώνεται περισσότερο πια στην ανάγκη να κλείσει το χάσμα μεταξύ έρευνα ε, και παραγωγής. Άρα θα τονώσει και αυτό την καινοτομία, εκεί επικεντρώνεται. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέσβη. Επόμενη ερώτηση από τον Σέλφο Σιλικιώτη από την ΚΟΕ. θα μιλήσω στη γλώσσα μου, ελληνικά. Κύριε Φερότζη, από το 2008 που ξέσπασε η οικονομική κρίση έχουν προωθηθεί πολλά μέτρα και υιοθετήθηκαν νέε πολιτικέ για στήριξη των τραπεζών, εν δεν έχουμε δει να γίνει το ίδιο για στήριξη τη βιομηχανία, τη πραγματική οικονομία και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ακούσαμε αρκετά από αυτά που είπετε, όμω δεν ακούσαμε μια νέα προσέγγιση, δηλαδή κίνητρα ανάπτυξη και εξειδικευμένα προγράμματα στήριξη και το πιο σημαντικό, απλοποίηση τη διαδικασία πρόσβαση ε, στη χρηματοδότηση ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το δεύτερο ερώτημα ε, από τη θέση σας ως πρόεδρος του International Affairs Institute of Rome αλλά και γενικότερα στο πλαίσιο της δράσης σας γνωρίζω ότι έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη συμφωνία TIP. Μπορείτε να μας πείτε και σε εσείς ίσως τις σημαντικότερες αρνητικές συνέπειες που θα υποστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την υπογραφή αυτής της συμφωνίας ε, και ιδιαίτερα πώς θα διασφαλιστεί ότι δεν θα πληγούν τα εργασιακά δικαιώματα και οι συλλογικές συμβάσεις. Ε, Κύριε Σιλικιώτη, ε, δεν κατάλαβα αυτό που αναφέρετε για τη συμφωνία. Ποια συμφωνία είπατε στο τέλος της παρέμβασής σας. TTIP. Uh, Ευχαριστώ για το ότι αναφέρετε πως ήμουν πρόεδρος του Ινστιτούτου Afar International παραιτήθηκα μόλις ορίστηκα ως υποψήφιος επίτροπος από την κυβέρνησή μου. Δεν είμαι πλέον, ενώσο είμαι επίτροπος τουλάχιστον. Για να, να απαντήσω στην ερώτησή σας, υπερβολική προσοχή στις τράπεζες, λιγότερη στην πραγματική οικονομία. Ναι, ίσως είναι μία από τις τακτικές κριτικές. Δεν είναι βέβαια αρμοδιότητά μου. Η Ένωση μεταξύ άλλων πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση στην, ε, ε στις, ε, σε χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Έχουμε ωστόσο τη δυνατότητα μέχρι, μέσω του προγράμματος COSME για την βοήθεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως ποσού ύψους 1,4 δις ειδικά για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πιστοτική υποστήριξη. Δεν είναι τεράστιο κονδύλι, είναι δεικτικό ωστόσο δείγμα της δέσμευση και υποστήριξης της Ευρώπης αυτού του συγκεκριμένου ε, τη προσέγγιση. Τώρα για το TTIP η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει πολλές ευκαιρίες, ανοίγει, την, διευκολύνει την πρόσβαση στην αμερικανική κυρίως αγορά που θα είναι θετική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Οι διαπραγματεύσεις είναι σύνθετες, το ξέρω. Η, το καθήκον μου για την περίοδο της θητείας μου είναι να επαγρυπνώ ούτω ώστε να εξασφαλίζω πως στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων οι αποφάσεις που λαμβάνονται δεν θα επηρεάσουν τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κυρίως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Επόμενη ερώτηση για τους πράσινους. Ο κύριος Πούτι Κόφελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς όρισατε κύριε Πρέσβη Νέλη Φερότσι. Χάρηκα που αναφέρατε ότι κατά τη γνώμη σας η ανταγωνιστικότητα και η εφορία δεν είναι ε, αντικρουόμενα, αλλά θα πρέπει να είναι αλληλοσυμπληρώμενα στοιχεία. Θα ήθελα να μάθω από εσά αυτό το πλαίσιο τι θα κάνετε βραχυπρόθεσμα για να βοηθήσετε να προωθηθούν δύο βασικές στρατηγικές που είναι η ενεργειακή αποδοτικότητα και η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων τα συγκεράσετε αυτά τα δύο. Και τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει πάντα βράχη πρόθεσμα για να δημιουργηθούν επενδύσεις. Γιατί ένα από τα μηνύματα που έστειλαν σε αυτό το κοινοβούλιο οι πολίτε στι τελευταίες εκλογέ, σύμφωνα με τη δική μου γνώμη πάντα, είναι ότι χρειαζόμαστε να αλλάξουμε από μια πολιτική που είναι στραμμένη στη λιτότητα και να πάμε ε, στις επενδύσεις. Όχι μακράς πνοής όμως ε, εξαγγελίες, βραχυπρόθεσμα και ένα πολύ σύντομο. Πολλοί εδώ στην Επιτροπή μας πιστεύουν ότι στο μέλλον η καινοτομία θα αποτελέσει και το κλειδί για τις εξελίξεις και τις επενδύσεις, αλλά θα πρέπει να είναι και πάλι στο χαρτοφυλάκιο της δικής σας αρμοδιότητας, της δικής σας γενική διεύθυνση επιχειρηματικότητας, DG Enterprise. Θα το φροντίσετε αυτό να επανέλθει για την επόμενη θητεία σε αυτό το χαρτοφυλάκι. Ευχαριστώ. Για το πρώτο σας ερώτημα, τα παραδείγματα που αναφέρατε είναι σημαντικά για την ενεργειακή απόδοση. Ο στόχος αυτός που θα οριστεί ίσως και την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η πρόταση της Κομισιόν θα βοηθήσει το συνδυασμό της βιωσιμότητας με την ανταγωνιστικότητα. Ένα τυπικό παράδειγμα μιας δέσμης μέτρων είναι αυτό που μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, μπορούν να μειώσουν ε, το κόστος και να τονώσουν την καινοτομία, ιδίω στον τομέα της οικοδομής, τον κατασκευαστικό κλάδο. Ταυτόχρονα μπορούν να συνεισφέρουν και στην ε, μείωση της ενεργειακής εξάρτησης. Ένα τυπικό παράδειγμα λοιπόν μιας δέσμης μέτρων τα οποία εάν ερμηνευτούν και εφαρμοστούν ορθά, δείχνουν ότι βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα είναι συμβατές έννοιες. Για τις επενδύσεις, μίζουν το ζήτημα, υπερβαίνει κατά πολύ τις ευθύνες ε, που με μεγάλη ταπεινότητα θα ασκήσω για λίγους μήνες, αλλά είναι κλειδί για την ε, επιτυχία της στρατηγικής μας για την ε, προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Ελπίζω με τις δικές μου δράσεις να έχουμε την, και με την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος Κόσμε ναι μεν περιορισμένα γιατί δεν έχουμε παραπεπερασμένα κονδύλια, να βελτιώσουμε κάπως την κατάσταση, να παράσχουμε εγγύσεις για δάνεια και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ΜΜΕ που επενδύουν για να διευρύνουν το πεδίο αρμοδιοτήτων τους, για να ε, αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους και εκτός εθνικών συνόρων. Είναι ένας στόχος λοιπόν ε, για την αύξηση των επενδύσεων στην Ευρώπη. Η καινοτομία στα πλαίσια της άμεσης ε, αρμοδιότητας γάμα δέλτα βιομηχανία επιχειρήσεις σε κάποιο βαθμό ναι ασκείται αυτή η αρμοδιότητα αλλά η διαχείριση ορισμένων συνιστοσών του προγράμματος ορίζον 2020 ήδη γίνεται, αλλά είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί εν τέλει από τον επόμενο πρόεδρο της Επιτροπής και από το επόμενο σώμα των Επιτρόπων. Εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να διατυπώσω συστάσεις. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος του EFDD, ο συνάδελφος Μπορέλη έχει το λόγο. Ε, θα μιλήσω Ιταλικά. Για να βγούμε από την φυστάμενη κρίση πιστεύω εξ να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής της Ένωσης και άλλους τομείς. Μιλήσατε για έρευνα και για κατάρτιση. Προφανώς χρειάζεται έρευνα για την καινοτομία και η δεύτερη για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων που υπενθυμίζω ότι περιλαμβάνουν ανθρώπους τους, τους τέσσερις αυτούς μήνες πιστεύετε μπορεί να φέσετε τις βάσεις για την μεγαλύτερη ανάπτυξη της έρευνας και την καλύτερη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων. Ναι, θα έλεγα. Διότι η έρευνα και η καινοτομία που συνδέονται στενά μεταξύ τους στον τρόπο λειτουργία στο πρόγραμμα πλαίσιο που είναι γνωστό ως Horizon 2020 είχε συνολική χρηματοδότηση 80 δις ευρώ. Δεν είναι ασήμαντος ασήμαντο το νούμερο αυτό, ιδίως όταν το συγκρίνουμε με τις δυνατότητες του προηγούμενου κύκλου χρηματοδότησης της έρευνας. Να προσθέσω επίσης ότι το ίμιση περίπου των 80 δις αφιερώνονται ειδικά στην έρευνα που συνδέεται με την παραγωγή. Την έρευνα που συνδέεται με την καινοτομία δηλαδή. Άρα είναι μια ανησυχία κοινή και ένα στόχος επί του οποίου και η τωρινή και σίγουρα η μελλοντική επιτροπή θα δεσμευτούν συγκεκριμένα ιδίω χρησιμοποιώντας το εργαλείο του Horizon 2020. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπονάνο, μία γεγραμμένος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξαιρετική παρέμβασή σας και ευχαριστώ γι' αυτό. Θέλω να μου απαντήσετε ωστόσο στις πολύ μικρές, για το θέμα των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Διότι πολλές μικρές επιχειρήσεις έχουν πολλές μικρές επιχειρήσεις είναι πολλές και έχουν κόσμο που δεν είναι αρκετό για την πρόσβαση σε πόρους. Είναι τόσο μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν πληροφορίες, ε, υφίστανται την υπερβολική γραφειοκρατία, δεν έχουν την δυνατότητα δηλαδή να πρόσβαση σε αυτά που τους διαθέτει η Ένωση. Τι πιστεύετε γι' αυτό. Μια παρατήρηση. Ε, λέτε όλοι ότι λύγεται σε τέσσερις μήνες, σαν το γιαούρτι. Αλλά υπάρχει γιαούρτι καλό και γιαούρτι κακό. Καλή τύχη. Θα προσπαθήσω να είμαι καλής ποιότητας γιαούρτι κύριε βουλευτά θέσατε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα υπογραμμίζοντας την ανάγκη να θέσουμε στη διάθεση των πολύ μικρών επιχειρήσεων πρόσβαση και στην ενημέρωση θεμελιώδες. Ήδη έχουμε ένα δίκτυο που είναι γνωστό ως European Enterprise Network EEN που συνεργάζεται με οργανώσεις και σε τοπικό επίπεδο επιμελητήρια, ανάλογες ε, τέτοιες δομές και που αποτελεί σημείο βασικής επαφής μέσω των οποίων οι μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη μπορεί να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στην ενημέρωση για τα ευρωπαϊκά κονδύλια που είναι στη διάθεση των μικρών επιχειρήσεων αλλά και για τις ευκαιρίες ε, επιχειρηματικού χαρακτήρα και προβολής τους προς τα έξω. Υπάρχει λοιπόν το εργαλείο, σίγουρα μπορεί να βελτιώσουμε τα πράγματα, να κάνουμε καλύτερες τις ε, γνώσεις των μικρών επιχειρήσεων. Τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουμε μια δημόσια διαβούλευση για την εφαρμογή την κατάσταση εφαρμογή και την βελτίωση του Small Business Act στο μέλλον. Αυτή η δημόσια διαβούλευση θα ήθελα να έχει και μεγάλη συμμετοχή η δημόσια διαβούλευση που θα γίνει βάσει ενό ε, εγγράφου της Επιτροπή που ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή εύχομαι να μας δώσει καλές ιδέες και προτάσεις βάσει των οποίων θα βελτιώσουμε το έργο της επιτροπή για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη. Τώρα βάσει των κανόνα Ντεόντ δύο συνάδελφοι από το ΕΛΚ και δύο από τους σοσιαλιστές θα έχουν το λόγο. Πρώτος ο συνάδελφος Ρούμπικ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είχα την εξής ερώτηση για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών που θα κυριαρχήσει στο μέλλον πιστεύω. Πώς μπορεί αυτή η βιομηχανία να συνεισφέρει στο στόχο του 20% της επαναβιομηχάνησης να επιτευχθεί και κυρίως τι γίνεται με την πρόσβαση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πώς θέλετε να τη δημιουργήσετε γιατί στα κράτη-μέλη ακριβώς ε, οι τηλεπικοινωνίες είναι αρκετά περιχαρακωμένες και κατακαιρματισμένες και δεν υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός. Εδώ ποιοι είναι οι στόχοι σας παρακαλώ. Uh, Mr. Κύριε Ρούμπιχ, όπως γνωρίζετε, είμαι περισσότερο αρμόδιος για ε, άλλα θέματα και όχι για τις τηλεπικοινωνίες που είναι αρμοδιότητα άλλου επιτρόπου. Βεβαίως γνωρίζω πόσο σημαντική είναι η ψηφιακή ατζέντα και η πλήρη υλοποίηση μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς ως εργαλείο ακριβώ για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Θα κάνω ό,τι μπορώ έτσι ώστε ο στόχος αυτός να υλοποιηθεί πλήρως και να ενταχθεί στο πρόγραμμα εργασιών και του της Επιτροπής αλλά και της επόμενης ή δυνατόν. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μια πρόταση απόφασης, ένα κανονισμός που πρότεινε η Κομισιόν, αλλά δέχτηκε και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για τη μείωση του κόστους της περιαγωγής, ε, το roaming, είναι ένα παράδειγμα ακριβώ πώς μπορούμε και σε ποιο βαθμό να επιτύχουμε μια πρωτοβουλία που είχε ως στόχο τη ρύθμιση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών μπορεί να τονώσει την ανταγωνιστικότητα. Ε, η μείωση του κόστους της περιαγωγής είναι καλή και για τον ιδιώτη καταναλωτή αλλά και για τις επιχειρήσεις οπωσδήποτε. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια σύνδεση που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και θα κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ για να το διατηρήσω στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. η κυρία Κομπούλα Νάτσι, πρώτη κυρία που θα μιλήσει τόσο αργά σε αυτή την προχωρημένη ώρα. Κάτι πρέπει να κάνουμε, δεν γίνεται να μιλάνε μόνο άντρες εδώ, να το αλλάξουμε αυτό. <laughs> well, the yours. Thank you on your... Ευχαριστώ πολύ. Μιλήσατε για τους πολίτες και την άποψη που έχουν ε, για την Ευρώπη, όπως είδαμε και με τις εκλογές, ότι η Ευρώπη είναι μακριά. Ε, επιχειρηματίες και επιχειρήσεις, ε, αυτοί τι πιστεύουν, πιστεύουν ότι η Ευρώπη κάνει το σωστό, Χάσαμε 3,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας ε, στον τομέα της, της μεταποίησης. Είπατε ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ε, ΜΜΕ, το κόσμο που αναφέρεται και αυτό ε, χρησιμοποιεί κονδύλια. Πολλές φορές όμως δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά κάποιες επιχειρήσεις. Άκουσα επίσης ότι οι οργανώσεις ε, ΜΜΕ δεν ε, συμμετείχαν. Ε, θα μπορούσατε ίσως αυτούς τους τρεις-τέσσερις μήνες να έρθετε σε επαφή με οργανώσεις ΜΜΕ ώστε να καταλάβουν ότι κάνει πράγματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η Ευρώπη και επίσης πώς μπορείτε να διευκολύνετε την διεθνοποίηση αυτών των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Να συμμετέχουν και αυτές σε προγράμματα για την έρευνα και την καινοτομία. 80, 80 εκατομμύρια, πολλά είναι τα χρήματα, αλλά μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά η μικρή επιχείρηση. Συμφωνώ μαζί σας. Το προανέφερα απαντώντας ερώτημα του κυρίου Μπονάνο ότι πολλές φορές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα να ενημερωθούν για το τι κάνει ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Άρα υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης της, ε, των επιδόσεων της ε, Κομισιόν σε ό,τι αφορά την ενημέρωση που παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και όπως είπα και για την λειτουργία του Ευρωπαϊκού Επιχειρηματικού Δικτύου, δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχει και ένα άλλο ε, εργαλείο αποτελεσματικό, δηλαδή το δίκτυο των ε, ΜΜΕ των απεσταλμένων των ΜΜΕ voice και στόχος αυτού του δικτύου είναι να παρέχουν στην Κομισιόν πληροφορίες για το τι θεωρούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσει των μεμονωμένων χωρών απαραίτητο να γίνει από πλευρά Κομισιόν και Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε δηλαδή να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στι μικρομεσαίες επιχειρήσει να συλλέγουμε τα παράπονά του, τα αιτήματά τους, ε, τι παρακλήσει του, Ό,τι αφορά τη διεθνοποίηση, ναι, κάνουμε κάποια πράγματα, θα κάνουμε ακόμη περισσότερα, ιδίω αξιοποιώντα ε, τα κονδύλια του προγράμματος COSME. Από τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ συνολικά είναι αυτή η πρικοδότηση του προγράμματος COSME. 900 εκατομμύρια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα χρησιμοποιηθεί αυτό το κεφάλαιο για τη στήριξη προγραμμάτων διεθνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Επόμενο ερώτημα, η κυρία Μπιρ Κούνεν. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Δύο Φινλανδές ε, και ρωτάμε και δύο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως είπατε κύριε Πρέσβη, οι μικρές, ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, θα διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία. Πολλέ φορέ όμω ασκείται κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί εκπονεί τις, όλα τα νομοθετήματα έχοντα υπόψη τι κυρίω τι μεγάλε επιχειρήσει οι ίδιες ε, νομοθετικές ρυθμίσεις ισχύουν για μικρές και για μεγάλες επιχειρήσεις και πολλές φορές οι μικρές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην γραφειοκρατία, στα όλο και περισσότερα νομοθετήματα που προωθούνται. Και αυτό βέβαια επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα. Κύριε Πρέσβη, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε αυτό το πρόβλημα ή τέλο πάντων θεωρείτε ότι είναι πρόβλημα ε, αυτός ο φόρτος από νομοθετήματα ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Απάντηση, ναι, αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα, το γνωρίζουμε, το έχουμε λάβει υπόψη. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συζητηθεί. Ανέφερα πριν το πρόγραμμα REFIT που έχει ως στόχο να δώσει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αναθεωρεί φυστάμενη νομοθεσία για να είναι λιγότερο δυσκίνητη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδίως ε, για αυτές που λόγω μεγέθους ουσιαστικά υπομίζονται και το μεγαλύτερο βάρος αυτών των υπερβολικών ρυθμίσεων. Προς δύο κατευθύνσεις θα κινηθεί η δράση μας. Προετοιμασία κατάρτιση νέας νομοθεσίας, όπου εκεί θα μελετήσουμε σημαντικά τον αντίκτυπο της νομοθεσίας για το κόστος που θα ε, συνεπάγεται η νέα νομοθεσία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεύτερον θα αναθεωρήσουμε την ήδη φυστάμενη νομοθεσία ούτω ώστε να γίνει, αν μπορώ να το πω έτσι, πιο, πιο φιλική προς τις ΜΜΕ. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα από τα πιο επίμαχα ε, νομοθετήματα σε ό,τι αφορά το κόστος ε, και τα βάρια της μικρομεσαίας επιχειρήσης είναι ο κανονισμός REACH Γνωρίζουμε ότι ο κανονισμός REACH που εγκρίθηκε εδώ και κάποιο καιρό είχε ως στόχο την εισαγωγή του συστήματος ε, καταχώρησης ε, για τις άδειες κυκλοφορίας χημικών προϊόντων. Διεξήγαμε μια ανάλυση του συστήματος αυτού ε, και είδαμε ότι σε ένα βαθμό αποδείχθηκε άκρος δυσκίνητο και πάρα πολύ μεγάλο βάρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό θέλουμε να προχωρήσουμε σε μια μερική αναθεώρηση του κανονισμού αυτού και για να μειώσουμε μεταξύ άλλων το διοικητικό φόρτο. Τι πρέπει να κάνουν δηλαδή μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την καταχώρηση αυτών των προϊόντων. Αυτό είναι ένα μόνο από τα πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τα υπερβολικά βάρη με, με τη νέα νομοθεσία που πέφτουν πάνω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό θα είναι κομμάτι και των δικών μου καθηκόντων αλλά και κατά πάσα πιθανότητα τη επόμενη επιτροπής. Τελευταία ερώτηση ο κ. Φαβαμάτο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε πρέσβη Φερνάντο Νελφερότσε, χαίρομαι που σας βλέπω εδώ. Ξέρω τη δουλειά που έχετε κάνει τα τελευταία χρόνια ως ε, μόνιμος αντιπρόσωπος Ιταλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαιρετική δουλειά κάνετε και είμαι βεβαισμένο και ότι σε τέσσερι μήνες θα πετύχετε πολλά. Το ερώτημά μου αφορά τον Χάλιβα. Τα τελευταία χρόνια μειώθηκε σημαντικά η ευρωπαϊκή σιδηρουργία. Είναι δεύτερος παραγωγός χάλιβα 11% ανά τον κόσμο, αλλά από την κρίση και μετά η παραγωγή του χάλιβα είχε μία μείωση κατά 27% σε σχέση με το επίπεδο πριν την κρίση. Χάθηκαν 40.000 θέσεις εργασίας στον τομέα. Εδώ προστίθεται και η σύμπτωση της εισόδου ε, εξωτερικών εξωευρωπαϊκών παραγωγών με μέσω ιδίως ε, ευνοϊκών συνεργασιών, κυρίως από Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία λοιπόν αντιμετωπίζει ταυτόχρονα μείωση της ζήτησης και αύξηση του όγκου πωλήσεων στην εσωτερική αγορά. Η ανακοίνωση της ε, για το πρόγραμμα δράσης για μια ευρωπαϊκή χαλιβουργία που θα είναι ανταγωνιστική και βιώσιμη στο πλαίσιο αυτό είναι ενδιαφέρουσα. Πώς θα ενθαρρύνεται την επίλυση της κρίσης στον κλάδο. Eh, eh, Κύριε Τζανονάτο, η Επιτροπή χάρη στο έργο του προκατόχου μου έχει ξεκινήσει από καιρό ένα πρόγραμμα δράσης για τον Χάλιβα με επίγνωση ότι ο Χάλιβας είναι ουσιώδη κλάδος για την διατήρηση της παραγωγής στην Ευρώπη. Παρότι υφίσταται έντονη πίεση λόγω ιδίως ε, του ανταγωνισμού, επιθετικού ανταγωνισμού από χώρες του τρίτου εκτός Ευρώπης με χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Να υπογραμμίσω κάποιες διαστάσεις του προγράμματος δράσης αυτού. Το πρώτο θέμα είναι, το είπαμε αλλά το επαναλαμβάνω γιατί είναι σημαντικό, είναι η πρόταση διατήρησης αμύωτου του καθεστώτος του λεγόμενου καθεστώτος carbon leakage, δηλαδή δωρεάν παραχώρηση ποσοστώσεων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα για, τον, για τις βιομηχανίες υψηλής ε, χρήσης ενέργειας, ιδίως της χαλιβουργίας. Ξεκινήσαμε και ήδη εν μέρη εισάγαμε σημαντική μείωση των ε, διοικητικών βαρών ε, που αντιμετωπίζουν οι χαλιβουργίες. Θα χρησιμοποιήσουμε, εν μέρη το κάναμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, πόρους από το Horizon 2020 για να ενθαρρύνουμε την έρευνα καινοτομίας με στόχο την εισαγωγή στην παραγωγική διαδικασία του χάλιβα τρόπους μείωσης του κόστους παραγωγής δραστηριοποιούμεθα σε διεθνέ επίπεδο για να εξασφαλίσουμε ένα ε, ε, ελάχιστο επισότιμο επίπεδο ανταγωνισμού με τους ετέ με τους ανταγωνιστές μας και έχουμε και κάποια εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε με κάποια επιτυχία για να εμποδίσουμε ε, εξαγωγές μέσω dumping των, των προϊόντων χαλιβουργικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρέζη. Θα ήθελα να σας ενημερώσω αγαπητοί συνάδελφοι ότι Η ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου μεταδίδει ε, απευθείας ε, την ε, συνεδρίασή μας στο διαδίκτυο. Κύριε Πρέσβη, τώρα θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε μια σύντομη καταληκτική τοποθέτηση. Πρόεδρε, νομίζω ότι θα μπορώ να είμαι πολύ σύντομος. Τελειώνω τις παρατηρήσεις μου με ευχαριστίες στους όλους τους βουλευτές που έλαβαν το λόγο και σας για τα σχόλιά σας, τα εισαγωγικά κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή τις ερωτήσεις. Οι περισσότερες ήταν οι εκφράσεις ειδικών ε, μελημάτων και ανησυχιών που οπωσδήποτε θα λάβω υπόψη ε, στη εργασία μου αν με επιβεβαιώσετε. Θα ήθελα επίσης να τονίσω και πάλι κάτι που είπα εισαγωγικά. Είμαι στη διάθεσή σας και παρακαλώ να με θεωρείτε στο πλευρό σας σε κάθε ευκαιρία για να οικοδομήσουμε πάρα πολύ επικοδομητικό διάλογο. Θεωρώ ότι η συνεισφορά του Κοινοβουλίου στη στρατηγική αυτή για την αναγέννηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας είναι εκ των ουκάνευ. Ήδη αυτό έχει αποδειχθεί στο πρόσφατο παρελθόν. Ανέφερα την έκθεση Beauty Coffer και νομίζω ότι θα συνεχίσει το Κοινοβούλιο να συνεισφέρει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανάγκη το Κοινοβούλιο και τη στενή και επικοδομητική συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς κύριε Πρέσβη. Και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από τις τρεις επιτροπές ε, που είναι εδώ παρόντες μαζί μας από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς, ε, Περιβάλλοντος και Μεταφορών. Θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο στην επόμενη ακρόαση ε, αντίστοιχη. Ευχαριστώ όλους τους συναδελφούς της Επιτροπής Ήτρε για τις ερωτήσεις και την υπομονή σας. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας αφιερώσατε και για τις απαντήσεις σας, για την προετοιμασία και φάνηκε νομίζω ξεκάθαρα ότι ήσασταν πάντα σε στενή συνεννόηση και συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο κύριο Αντώνιο Ταγιάννη, πράγμα που ε, μας βοηθάει όλους. Ευχαριστώ πολύ. Δέκα λεπτά διάλειμμα και στη συνέχεια συνεδριάζουν οι συντονιστές. Δέκα λεπτά διάλειμμα η Επιτροπή στις Βρυξέλλες την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα συνεδρίασε της Επιτροπής που θα είναι η δεύτερη τακτική συνεδρίαση. Ευχαριστώ.